presidente la seduta è ripresa. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση μας. Ανακοινώ τα αποτελέσματα του δευτέρου γύρου των ψηφοφοριών για εκλογές αντιπρόεδρων. Αριθμός ε, ψηφισάντων 672. Λευκές ή άκυρα, λευκά άκυρα 34. ...638 ψήφοι... ...απόλυτη πλειοψηφία... ...320. Σας διαβάζω τις ψήφους που πήραν οι διάφοροι υποψήφοι. Κύριος Λάμστορφ, 393 ψήφοι. Λούνατσεκ, 441 ψήφοι. Ο κ. Παδημούλης, 469 ψήφοι. Πάσκου, 517 ψήφοι. Τάραντ. 261 ψήφοι. Εκλέγονται κύριοι Πάσκου, Παπαδημούλης, Λούνατσεκ και Λάμπτερτ. Πέτυχαν την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων. Και βάσει του δεύτερου γύρου έχουν εκλεγεί αντιπροέδροι του Κοινοβουλίου και τους συγχαίρω θερμά τους συναδέλφους αυτούς για το επιτευχθέν αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τα άρθρο 17, παράγραφος 2 του κανονισμού, λοιπόν η σειρά προτεραιότητας των αντιπροέδρων καθορίζεται από τη σειρά σύμφωνα με την οποία αυτοί έχουν εκλεγεί και σε περίπτωση ισοψηφίας από την ηλικία. Η συνθεσία του Προεδρείου θα κοινοποιηθεί στους Προέδρους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, όσον αφορά την εκλογή των κοσμητόρων, προτείνω να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιωτήτων στις 16 ώρα 4 το απόγευμα. Πρέπει να κατεθούν υποψηφιότητες στην Γενική Γραμματεία ε, στο R00101, στο γραφείο R00101 το, το ανοιχτό χώρο, το open space Προεδρία στο Louis Weiss. Ο πρώτος γύρος ψηφοφοριών θα ξεκινήσει στις 16.30 για την εκλογή κοσμήτωρων. Τα πρακτικά της θεσινής συνεδρίασης έχουν διανεμηθεί, υπάρχουν παρατηρήσεις.